θα έχω, είχα μια ανακοίνωση πριν περάσουμε στην επόμενη συζήτηση να σας πληροφορήσω ότι βάσει το άρθρο 231 εδάφιο 4 δεν υπήρξε έτοιμα να ψηφιστεί το διορθωτικό που ε, αναγγέλθηκε χθες τις 5 Οπότε θεωρείται εγκεκριμένο το διορθωτικό αυτό. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα στην εμμερήσια διάταξη.